και ελπίζουμε να επιστρέψει η ανάπτυξη και η ευημερία στην Ιρλανδία το ταχύτερο δυνατόν χάρη σε αυτά τα μέτρα. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πέρα τη συζήτηση. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι η κατάσταση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος σε θέματα ασύλου μετά την τελευταία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το το λόγο έχει η κυρία Μάλστρομ, την οποία και χαιρετίζω θερμά. Σας έδωσα το λόγο κυρία Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, η απόφαση της 21ης Ιανουαρίου του ΕΔΑΔ στην υπόθεση της Ελλάδας και του Βελγίου δείχνει ότι θα πρέπει να ορίσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να προβάλλουν επαρκή προστασία μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού και εκτιμένου και του κανονισμού του ε, Δουβλίνου τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να απαλλαχθούν ποτέ από την υποχρέωσή τους να προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτή την απόφαση το ΕΔΑΔ ορίζει και επαναλαμβάνει αυτή την αρχή. Βεβαίως δεν ορίζει το πώς θα λειτουργεί ο κανονισμός του Δουβλίνου. Θα πρέπει όμως να έχουμε ένα σαφές σύστημα για να δούμε ποιος θα ορίσει και θα χορηγήσει το άσυλο, ποιος θα ε, προσδιορίσει ότι κάποιος είναι ε, πρόσφυγας και πώς θα ορίσει την κατάσταση σε σχέση με πολλαπλές αιτήσει. Η αξιολόγηση όμως του κανονισμού του Δουβλίνου δείχνει ότι υπάρχει χώρος μεταρρύθμισης. Ήδη το 2008 είχαμε διαπιστώσει χάσματα και προσπαθήσαμε να τα αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα, τα αιτήματα, μάλλον τις αιτήσει των ενδιαφερομένων. Χαίρομαι για την υποστήριξη από το Κοινοβούλιο της πρότασης της Κομισιόν και θα ήθελα να συνεργαστούμε έτσι ώστε να φτάσουμε σε έναν πολύ σωστό κανονισμό του Δουβλίνου, κανονισμό υπαριθμών 2. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αναστολή μεταφορών σε περίπτωση που υπάρχει πίεση από πλευράς της πρώτης χώρας χορήγησης ε, ασύλου ή υποδοχής. Γιατί μέχρι τώρα υπάρχει διακριτική ευχέρεια έτσι ώστε να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των εταίρων του Δουβλίνου η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλη πίεση εξαιτίας των μεγάλων ροών μεταναστών στο έδαφος της και είναι δύσκολο να λειτουργήσει σωστά το σύστημα χορήγησης ασύλου στη χώρα αυτή. Εμείς το Νοέμβριο του 2009 είχαμε κινήσει μια διαδικασία επί παραλήψη κατά της Ελλάδας. Η Ελλάδα τόνισε ότι θα μεταρρυθμίσει το σύστημα χορήγησης ασύλου με βάση ένα πρόγραμμα δράσης που υποβλήθηκε στην Κομισιόν πέρσι το καλοκαίρι και έκτοτε έχει λάβει χώρα ένα νομοθετικό έργο στην Ελλάδα. Επίσης, καταβάλουμε προσπάθειες βοήθειας, χορήγησης βοήθειας προς την Ελλάδα και προβάλλουμε πρακτική και οικονομική αρρωγή για την ε, διαχείριση των συνόρων και καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και σχέσεων με τις γείτονες χώρες, ιδιαίτερα την Τουρκία. Άρα θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι βασιζόμαστε στη δημοκρατία, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην ισότητα και στο κράτος δικαίου, καθώς και την τήρηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε το δικαίωμα του ασύλου και θα συνεργαστούμε για μία πραγματική πολιτική χορήγησης ασύλου έτσι ώστε να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Βέμπερ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η πολιτική των προσφύγων έχει μεγάλη επικαιρότητα. Το βλέπουμε και στην Λαμπεντούζα, το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Και συγκινεί τους πολίτες της Ευρώπης. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι, πιστεύω, διότι έχουμε επιτύχει υψηλέ προδιαγραφέ για την προστασία των προσφύγων στην Ευρώπη. Έχουμε αναπτύξει προδιαγραφέ υψηλέ και για το πώ θα χειριστούμε ζητήματα παιδιών ή οικογενειών. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τι προδιαγραφέ μα αυτέ και η Ευρώπη είναι ένα χώρο θαλπορή για του ταλαιπωρημένου ανθρώπου αυτού του κόσμου. Αυτό όμω ταυτόχρονα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο στις δηλώσεις, αλλά πρέπει να προχωρούμε και σε δράση. Από τις δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του Βελγίου και από τη δικαστική απόφαση βάρος του Βελγίου και της Ελλάδας βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί ικανοποιητικά το σύστημα στην πράξη. Και γι' αυτό η Επιτροπή μαζί με τα προγράμματα δράσης θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, ώστε γρήγορα να είμαστε σε θέση να ε, τηρούμε στην ουσία τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδος θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε σύνορα που μπορούμε να διασφαλίσουμε και από τις δύο πλευρές και αισθάνομαι μεγάλη απογοήτευση για τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία ως εταίρος χώρα συμπεριφέρεται. Δεν έχει ακόμα συναυτή συμφωνία επαναπροώθησης με την Τουρκία. Ε, πράγμα το οποίο είναι υποχρέωση της Τουρκίας εφόσον θέλει να καταστεί μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό καλώ την Τουρκία από αυτή τη θέση να προβεί σε ισχυρότερες προσπάθειες, σαφέστερες προσπάθειες για την υπόθεση αυτή. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Ταμείο για τους Πρόσφυγες με η Frontex, συγκεκριμένη πρακτική βοήθεια μπορούν να αποτελέσουν τρόπου στήριξης της Ελλάδας στην περίπτωση αυτή των συνόρων της αλλά και της Λαμπεντούσας για την Ιταλία. Ζήτημα αλληλεγγύης δεν τίθεται για μας. Είναι τώρα η ώρα να προσφερθεί αυτή η αλληλεγγύη. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βέμπερ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Λαμπρινίδης. Μινούτο. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, όπως ανέδειξε η απόφαση του δικαστηρίου, είμαστε όλοι παγιδευμένοι στο Δουβλίνο 2. Ως αποτέλεσμα της ανισοκαταμερούς κατανομής των βαρών εδώ, έχουμε τα κράτη-μέλη σε ένα πινκ-πονγκ ευθυνών και καταγγελιών εδώ και χρόνια, με τους ατυχείς πρόσφυγες εγκλωβισμένους στη μέση. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελευταία χρόνο η Ελλάδα έχει υποδεχτεί 90% μεταναστών και ετούντων άσυλο στην Ευρώπη τώρα με την αλγερία η πίεση μεταφέρεται στην ιταλία. ω πότε κάποιοι θα επιμένουν να προσποιούνται ότι αυτό είναι ελληνικό ιταλικό μαλτέζικο κυπριακό πρόβλημα. τα σύνορα των χωρών μα είναι σύνορα ευρωπαϊκά. η αναπτυξιακή μα πολιτική η εξωτερική μα πολιτική ή η έλλειψή του είναι ζητήματα ευρωπαϊκά. με τη στεναρή συνδρομή τη ευρωπαϊκή επιτροπή η χώρα μου έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο τεράστια βήματα για τη βελτίωση τη κατάσταση του αλλά αυτό προφανώ δεν αρκεί πρέπει το νέο δουβλίνο να σταματήσει τις μαζικές επιστροφές στο πρώτο κράτος μέλος πρέπει να εγκαθιδρύσει μια πραγματική ουσιαστική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. αυτό το έχει ζητήσει το κοινοβούλιο. ήρθε ο καιρός πια κάποια κράτη στο συμβούλιο να σταματήσουν να παίζουν τους πόντιους πιλάτες και να σνίπτουν τα σχήρες τους. ευχαριστώ η κυρία Βίκστρομ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δείχνει σαφέστατα ότι παραβιάστηκαν τα άρθρα 3 και 13 της ε, Σύμβασης από την Ελλάδα και το Βέλγιο. Ε, απαξιωτική ε, ταπεινωτική συμπεριφορά ενός Αυγανού μετανάστη που πήγε από την Ελλάδα στο Βέλγιο. Αυτή είναι η περίπτωση και ακολούθησε η απόφαση που φυσικά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ε, ο εισηγητής για την αναθεώρηση του κανονισμού Δουβλίνου 2 καλωσόρισε την απόφαση του δικαστηρίου διότι καταδεικνύει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διακόψουν ε, τις ε, μεταφορές προς την Ελλάδα όσο δεν τροποποιούνται αυτές οι πρακτικές. Επίσης, καταδεικνύεται ότι υπάρχει και μια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε μέχρι το 2010 ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, λέμε ωραία, αλλά θα πρέπει να βοηθούμε ένα για να το πετύχουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αλλάξει τη στάση της για το Δουβλίνο 2, γιατί είναι ο ακρογωνίος λίθος της ε, κοινή πολιτικής ασύλου. Επίσης υπάρχουν στατιστικά ε, στοιχεία που δείχνουν προς ποια κράτη-μέλη θα πρέπει να γίνονται οι επιστροφές. Επίσης υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές περιπτώσεις που πρέπει να εξεταστούν. Το Κοινοβούλιο έχει σαφέστατη θέση για το Δουβλίνο 2 και αναμένει τις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις. Ναρωτιόμαστε λοιπόν τι θα γίνει με το μηχανισμό αλληλεγγύης, με τα δικαιώματα των ανηλίκων και τα ένδικα μέσα. Σημαντικά στοιχεία του Δουβλίνου, του Δουβλίνου 2. ελπίζουμε να συνεχίσουμε την αγαστή συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμή. Σας ευχαριστούμε. Τώρα, ε, για δύο λεπτά από τους πράσινους. Το ζήτημα είναι ότι τι θα κάνουμε τώρα, τι πρέπει να γίνει τώρα τη στιγμή που αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όρισε ότι οι ετούντες άσυλο δεν πρέπει να μεταφουν στην Ελλάδα. Ελέγχθη ότι θα βοηθήσουμε την Ελλάδα έτσι ώστε να μπορέσει να ορίζει καλύτερα και να διαχειρίζεται καλύτερα τα σύνορά της και δεν θα στείλουμε μετανάστες πίσω στην Ελλάδα με βάση τον κανονισμό του Δουβλίνου. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι πάντα αυτή η σωστή ε, απάντηση. θα πρέπει να υπάρχει μία ρήτρα αλληλεγγύης με βάση το σύστημα του Δουβλίνου. Διαφορετικά θα υπάρχει ανισομερής μεταχείριση. Με βάση και τη δική μου χώρα, στη Βόρειο Θάλασσα, δεν έχουμε ε, σωρία μεταναστών που φτάνουν στην Ολλανδία με αυτοσχέδια σκάφη, με σχεδίες στην ουσία. Θα πρέπει όμως πάντα να αναμένουμε ενδεχόμενους κλειδονισμούς. Συμφωνείτε ότι το σύστημα του Δουβλίνου στην ουσία έχει περιπέσει σε αχρηστία. Πότε μπορούμε να το αναθεωρήσουμε νομίζετε και πιστεύετε ότι οι βόρειες χώρες θα πρέπει να καταδείξουν αλληλεγγύη πλέον θα ήθελα τη γνωμοδότησή σας ως προς την απόφαση του ΕΔΑΔ την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές. Έχουμε μία αύξηση φόρτου εργασίας κατά 4.000% διότι είδαμε ότι το σύστημα του Δουβλίνου δεν είναι λειτουργικό. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλος φόρτος εκκρεμών υποθέσεων. Νομίζω ότι η βελγική κυβέρνηση θα πρέπει να καταβάλει το μεγαλύτερο αντίτιμο, διότι η βελγική κυβέρνηση αμέλησε να ανταποκριθεί. Πότε θα βελτιωθεί ε, το σύστημα του Δουβλίνου, έτσι ώστε να μην υπάρχει τόσο απάνθρωπο σύστημα. Κυρία Σαρτζεντίνη, με βάζει την ε, μπλε κάρτα, θέλει ε, κάποιος να σας ε, απευθύνει ένα ερώτημα. Μπορείτε να το δεχτείτε. Έχετε το λόγο. Κυρία Σαρτζεντίνη, γιατί δεν λέτε ότι η Τουρκία έχει απόλυτο, έχει μεγάλο λάθος όταν αποστέλει όλους αυτούς τους μετανάστες στην Ελλάδα. Γιατί λέτε ότι καταχρώμεθα το σύστημα ασύλου. Γιατί δεν μιλάτε για λαθρομετανάστες και εγκληματίες οι οποίοι στην ουσία καταχρώνται το σύστημά μας. Μπορείτε να απαντήσετε. Η κυρία ε, Σαρτζεντίνη. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω στον κύριο Μαντλένερ. Νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να εξετάζει τη δική του συνείδηση. Η Ευρώπη θα πρέπει να βελτιώσει το δικό της σύστημα και να βοηθήσει την Ελλάδα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις περιπτώσεις των ετούντων άσυλο πριν κινηθεί εκτός των συνόρων της. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε λοιπόν εντός των δικών μας συνόρων. Συμφωνώ κύριε Μαντλέρα ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τους ε, λάθρομετανάστες και τους ε, ε, εμπόρους και οπωσδήποτε θα πρέπει να δούμε πώς και η Τουρκία αντιμετωπίζει το θέμα των μεταναστών που προέρχονται από αλλού. Αλλά ας δούμε τις δικές μας ευθύνες καταρχήν και μετά ας επεκταθούμε στους άλλους. Ο κύριος Κύρκο, πια 1,5 λεπτό καθίσταται σαφές ότι μιλάμε, με ένα, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί πλέον και δυστυχώς το νομοθετικό σκέλος και το εκτελεστικό βρίσκονται σε κατάσταση ρήξης και μιλάμε για μια νέα ερμηνεία του νόμου. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με βάση ένα νέο σύστημα το οποίο δεν θα είναι δικτατορικό. Δηλαδή δεν θα μιλάμε για αποφάσεις δικαστηρίων, αλλά μέσω αλληλεγγύης και καλής επικοινωνίας μεταξύ γειτόνων χωρών θα αντιμετωπίσουμε τον φόρτο αυτό, διότι ο φόρτος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μετατοπίζεται σε άλλα κράτη-μέλη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι αποζητούν μία ε, ελεύθερη ζωή αλλά η πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΔ μιλά για την ευρωπαϊκή νομοθεσία εντός ε, κρατών μελών, σε επίπεδο κρατών μελών. Θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση μακροχρόνια και μπορείτε να μας πείτε ότι δεν θα δημιουργήσουμε επιπρόσθετη νομοθεσία η οποία κάποια στιγμή θα ανατραπεί από ένα μελλοντικό δικαστήριο πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την Ελλάδα και άλλα κράτη-μέλη που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν έναν τόσο μεγάλο φόρτο. Ευχαριστούμε κύριο Κίρκοπ. Ο κύριος Ντε για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Επιτροπή κυρία Μάρστρομ η οποία πήθηνε την προηγούμενη εβδομάδα έκκληση στα κράτη-μέλη να ασχοληθούν με το θέμα του ασύλου και πρόκειται για ένα θέμα ακανθόδες. Όμως οι μεγάλες ροέ προσφύγων από την Τινησία αποδεικνύουν τις δυσκολίε που έχει η, η Ιταλία ως προς την αντιμετώπιση αυτών των ροών και εάν τα λοιπά κράτη της Ευρώπης μείνουν με σταυρωμένα χέρια θα είναι αδύνατο για την Ιταλία μόνη της να αντιμετωπίσει αυτές τις ροές. Πρέπει λοιπόν κατεπηγόντως, όπως άλλωστε προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αναλάβουν δράση ε, στο πλαίσιο της συνθήκης του Βλήνου και σε, μέσα από μια συμφωνία δεσμευτική για τις διαδικασίες του ασύλου τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει εάν βλέπει κάποιο τρόπο εμείς να της προσφέρουμε υποστήριξη ώστε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεγιόγκ. Το λόγο έχει ο κύριος Μάντλερ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι κάτω για άλλη μια φορά και αφού η Ευρώπη έχει στηρίξει με δισεκατομμύρια την Ελλάδα για να ε, ξεφύγει από την κρίση, έρχεται τώρα ή καλείται τώρα να προσφέρει χείρα βοηθείας για το θέμα των προσφύγων. Εμείς ε, υποφέρουμε διαρκώς και βλέπουμε μπροστά μας συνέχεια τα προβλήματα της υποτιθέμενης πολιτισμικότητας και της ανύπαρκτης ενσωμάτωσης. Τέτοιου είδους φόρτο βάρος, άχθο δεν θέλουμε. Πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική πολιτική ασύλου στην Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει πέσει θύμα του κακού της γείτονα, της Τουρκίας και θα πρέπει να την στηρίξουμε. Η Ελλάδα πρέπει να χτίσει το τείχος που θα εμποδίσει αυτούς τους μετανάστες που έρχονται από την Τουρκία και τις μεγάλες ροές προς την Ελλάδα. Πρέπει να χτιστεί το τείχος και πρέπει να τιμωρηθεί η Τουρκία η οποία επιτρέπει σε αυτές τις μεταναστευτικές ροές, αυτούς τους λάθρο μετανάστες να περνούν τα σύνορά της η πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γίνει πολύ πιο αυστηρή και άτεγκτη. Είναι τεράστιο το ποσοστό των ετούντων το άσυλο που δεν είναι πραγματικοί ε, πρόσφυγες αλλά μόνο ε, άνθρωποι που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις καταστάσεις. Ο κ. Παπα-Νικολάου. Θα κάνω μία υπόθεση. Βλέπουμε την αναταραχή που υπάρχει στις χώρες της Μεσογείου και στις χώρες του αραβικού κόσμου. Βλέπουμε ότι πολλοί πολίτες των χωρών αυτών επιδιώκουν να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στην ευρώπη. ήδη αυτό είναι μια πραγματικότητα και φοβάμαι ότι και η υπόθεση που θα αναπτύξω και αυτή μπορεί σύντομα να είναι πραγματικότητα. έρχονται λοιπόν οι πολίτες των τρίτων αυτών χωρών στην ευρώπη. φτάνουν στην λαμπεντούζα βλέπουμε εκεί τα προβλήματα κάποιοι άλλοι προσπαθούν μέσω της τουρκίας να φτάσουν στην ελλάδα και αξιοποιούν τη δυνατότητα να μην αιτούνται για βίζα με βάση τις συμφωνίες που έχουν οι τρίτες χώρες αυτές με την τουρκία πολλές από αυτές κάποιοι άλλοι πηγαίνουν στη μάλτα κάποιοι άλλοι ενδεχομένως στην πορτογαλία και την ισπανία. στη συνέχεια κάποιοι από αυτούς αιτούνται άσυλο. είναι δεδομένο ότι εκεί θα έχουμε πάλι εφαρμογή του δουβλίνου 2. και ξέρετε αν και τότε υπάρξει προσφυγή κάποιου ε, ετούντα άσυλο για τα θέματα αυτά και πάλι θα υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις όπως και μέχρι σήμερα είχαμε καταδικαστικές αποφάσεις από εθνικά δικαστήρια πριν φτάσουμε στην απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου. ας μην υποκρινόμαστε λοιπόν. και κάτι ακόμα υπάρχουν κάποιοι που θα συλληφθούν και δεν θα δικαιούνται άσυλο. ξέρετε με βάση τη συμφωνία την οποία το πέρας των διαπραγματεύσεων ανακοίνωσε η επιτροπή για να όσοι μπουν από την τουρκία για να επιστραφούν με επανεισδοχή στην τουρκία θα πρέπει να περιμένουμε δύο χρόνια για να εφαρμοστεί η συμφωνία και τρία χρόνια που είναι η μεταβατική περίοδο για του υπηκόου τρίτων χωρών πέντε χρόνια. Αυτού δηλαδή που θα συλλάβουμε αυτή την περίοδο με βάση την κρίση που αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να περιμένουμε το 2016 ή το 2017 για να του δεχτεί πίσω η τουρκία. επιτρέψτε μου να πω ότι με τέτοια διαχείριση πολύ φοβάμαι ότι η ευρώπη δεν στέκεται σήμερα στο ύψο των περιστάσεων. Η κυρία Σιλβίγκη Γιόμ ε, τώρα για δύο, λεπ... για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, νομίζω είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε διάφορε δεσμεύσει. Σε Οκτώβριο 2008, ε, το σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Είπαμε τότε ότι ήρθε η ώρα να αναλάβουμε πρωτοβουλίε, ούτω ώστε να επισπευτεί η συγκρότηση ενό ευρωπαϊκού συστήματο ασύλου και να κατοχυρώσουμε μια αποτελεσματικότερη προστασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο χρόνια μετά την υπόσχεση αυτή, έχουμε τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναχείρα, αλλά διαπιστώνουμε ότι η όλη διαδικασία ε, ε, θέσπιση του κοινού συστήματος ασύλου ε, καθυστερούν. Ε, ε, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Βλέπουμε τις ατέλειες με την τελευταία απόφαση του ελληνικού συστήματος, αλλά με την απόφαση περνάει ένα σαφέ μήνυμα, ενώ η Ελλάδα τροποποιεί το εθνικό τη σύστημα και την ενθαρρύνει να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες. Τώρα, ας περάσω σε ένα γενικότερο θέμα. Το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, ένα από τα θεμέλια, η νέο κανονισμός ε, Δουβλίνο και το βασικό αξίωμα ότι ε, ισχύουν οι ίδιοι όροι για το άσυλο μέσα στην Ένωση. Έχει δημιουργηθεί μία ανισότητα με το τωρινό σύστημα και για τους ετούντες άσυλο αλλά και για τα ίδια τα κράτη-μέλη γιατί δεν εφαρμόζονται οι ίδιοι όροι αναμένοντας ένα λειτουργικό ελληνικό σύστημα ασύλου αναβάλλονται οι αιτήσει προς την Ελλάδα ε, και δεν αναλαμβάνεται η εξέταση των φακέλων. Επίσης, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στέλνει ένα μήνυμα και προς όλους τους υπόλοιπους ε, ε, συναρμόδιους φορείς. Χρειάζεται μεταρρύθμιση του συστήματος, κυρίως του κανονισμού Δουβλίνο. Ε, σας μίλησα για την αναβολή των μεταβιβάσεων που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, ρίχνει νέο φως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σε αυτόν τον μηχανισμό και στην Ευρωπαϊκή συνεργασία για τα θέματα ασύλου και προκύπτει ότι χρειαζόμαστε τη θέσπιση ενός τέτοιου μηχανισμού αναβολής παγώματος Επίσης, ε, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων υπάρχουν και άλλες τροποποιήσεις που έχουν υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τον τωρινό κανονισμό, κυρίως παραδείγματος χάρη σε σχέση με τις εγγυήσεις που συνδέονται με αυτό το μηχανισμό. Τέλος, ε, χάρη στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μπορούμε να αρχίσουμε και τη συζήτηση για τους ετούντες άσυλο και την επισφαλή τους ε, θέση, ούτω ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν προσφυγή αν κρίνουν ότι υπάρχει παραβίαση κατά την εφαρμογή του κανονισμού Δουμπλίνο. Ε, όλοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καταδεικνύεται ότι ε, χρειαζόμαστε ένα νέο υπεύθυνο σύστημα ε, ασύλου. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Χίρς τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, σήμερα ε, συζητούμε το θέμα της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ουσιαστικά δεν εξετάζουμε μόνο το θέμα του Βελγίου, γιατί και η Γερμανία αποφάσισε να μην επαναπέμπει τους ετούντες άσυλο στην Ελλάδα, να παγώσει τη διαδικασία μέχρι νεοτέρας. Τίθεται λοιπόν ε, το ζήτημα όπως ακριβώς μας το περιέγραψαν οι συνάδελφοι να φτιάξουμε ένα τείχο παραδείγματος χάρη που θα περιβάλλει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να λύσουμε το πρόβλημα ή και φυσικά εμείς αυτή τη λύση προκρίνουμε ε, να προστατεύσουμε του ετούντες άσυλο ε, βάσει ενό πιο οργανωμένου συστήματος. Αυτό όμω σημαίνει ότι ο ετών άσυλο θα έχει την, στη διάθεσή του έναν μηχανισμό που λειτουργεί εύρυθμα για να λειτουργήσει όμως εύρυθμα χρειάζεται ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν είναι επιτρεπτό κάποια κράτη-μέλη να υπομίζονται όλη την ευθύνη. Ε, ας λάβουμε υπόψη τη γεωγραφική θέση κάποιας ε, χώρας. Είναι λογικό ότι κάποιες χώρες έχουν ένα ισχυρότερο ρεύμα μεταναστών. Δείτε τι γίνεται ε, με τους μετανάστες από την, Ισία στη Λαμπεντούζα. Είναι δυσβάσταχτη κατάσταση. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ένα κράτος μέλο. Επίσης να σας θυμίσω ότι είχε γίνει με το κοσυφοπέδιο. Άλλο κύμα μεταναστών. Και εμεί βρεθήκαμε, μα κατέλαβε εξαπίνηση η εξέλιξη και δεν μπορέσαμε, αν θέλετε, να διαχειριστούμε ε, αυτή την αυξημένη ροή μεταναστών. Ε, λοιπόν, για να βελτιώσουμε τον κανονισμό Δουβλίνο 2, δεν αρκεί αναθεώρηση. Χρειάζεται μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Σα ευχαριστούμε. Ε, Κυρία Κάρμεν Ρομέρο Λόπες για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Όπως ξέρετε, η απόφαση του ΕΔΑΘ δεν βασίστηκε σε έναν Αυγανό, ο οποίος ήταν ε, αντικείμενο εμπορίου, αποτέλεσε αντικείμενο ε, δουλείας. Είχε αιτηθεί άσυλο και χρειαζόταν ε, διεθνή προστασία. Η απόφαση έχει σημασία με βάση το περιεχόμενο, διότι θα πρέπει να, να μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος αυτός μπόρεσε να προσφύγει, άλλοι δεν μπορούν. Θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί σε σχέση με το ΕΔΑΔ και τα κράτη-μέλη. Μας ενδιαφέρουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ζητούμε από τους ετούντες να μην βρίσκονται σε αυτή την επώδυνη κατάσταση. Δυστυχώς όμως οι πρόσφυγες βρίσκονται σε κέντρα κράτησης ή συγκέντρωσης κάτω από απάνθρωπες συνθήκες αναμένοντας την έκβαση της αίτησης και, όλες οι... και δεν ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες σε όλα τα κράτη-μέλη. Δυστυχώς υπάρχει έλλειψη αλληλεγγύης, γι' αυτό ζούμε αυτές τις ε, καταστάσεις. Μιλάμε για αποζημίωση, για ηθική βλάβη. Τι αποζημιώσεις ε, μπορούν να ζητήσουν όμως αυτοί οι άνθρωποι τη στιγμή που υπόκεινται κατά σε κέντρα συγκέντρωσης. Νομίζω ότι χρειάζονται πολύ περισσότερο από τον κανονισμό του ε, Δουβλίνου και θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρηγορότερα και επί της ουσίας. Ευχαριστούμε. Κύριε Βίσπεκ, θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα της μπλε κάρτας ή θέλετε να ενταχθείτε στη διαδικασία Catch the Eye. Ωραία, την άλλη φορά να, το, να επιδείξετε την μπλε σας κάρτα, παρακαλώ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Μπουζούτιλ. Η ε, απόφαση του ΕΔΑΔ δεν αφορά μία απόφαση κατά του Βελγίου ή της Ελλάδας καταφέρεται κατά του κανονισμού του Δουβλίνου, διότι ο κανονισμός του Δουβλίνου επέτρεψε στο Βέλγιο να μεταφέρει τον Αφγανό πολίτη εκ νέου στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό οι παραμεθόριες χώρες να είναι αυτές που να αναλαμβάνουν ολόκληρη την ευθύνη και το φόρτο εξ ολοκλήρου, διότι οι χώρες αυτές δεν είναι οι θεματοφύλακες ή δεν αποτελούν δεν μπορούν να ε, επιτελέσουν ρόλο αστυνόμευσης για όλα τα κράτη-μέλη. Άρα όταν μια χώρα μεταφέρει τους ετούντες άσυλο σε μια άλλη χώρα που βρίσκονται υποπίεση όπως η Ελλάδα εκείνο το χρονικό διάστημα, αυτό σημαίνει παραβίαση ανθρωπίνων και δωμάτων και παραβίαση της χάρτας. Αυτό το αναγνώρισε η Γερμανία και έχει αναστείλει τις μεταφορές ε, ετούντων προς την Ελλάδα. Θα πρέπει όμως να αναμορφωθεί ο κανονισμός του Δουβλίνου το ταχύτερο δυνατόν. Ο κύριος Μαυρονικόλας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ο λόγος για τον οποίο νιώθω την ανάγκη να μιλήσω στη σημερινή συνεδρία είναι ακριβώς διότι δεν έχει αναφερθεί το θέμα της κύπρου και το πρόβλημα της μετανάστευσης που αντιμετωπίζουμε. η κύπρος ένα μικρό κράτος του μισού εκατομμυρίου δέχεται καθημερινώς εισδοχή μεταναστών μέσω των κατεχομένων περιοχών περνώντας την πράσινη γραμμή σε έναν αριθμό που μπορεί να φτάνει και τους 30 με 50 άτομα ημερησίως σε έναν πληθυσμό μισού εκατομμυρίου. Εμείς δεν διαθέτουμε κέντρα συγκέντρωσης των αιτητών ασύλου και αποτέλεσμα τούτου οι αιτούντες πολιτικών άσυλων δεν μπορούμε στο τέλος της ημέρας εάν δεν γίνει αποδεκτή η αίτησή τους να τους στείλουμε πίσω στην χώρα από την οποία προέρχονται. εισέρχονται από τα κατεχόμενα πλήστες των φορών καταστρέφουν τα έγγραφά τους και ουσιαστικά οι μετανάστες αυτοί παραμένουν στο νησί. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαυρονικόλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Όντως, τα θέματα του ασύλου, τα προβλήματα δεν λύνονται με τύχη. Και γι' αυτό ήθελα να πω ότι όποιος καλεί για χτίσιμο τυχών δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να μείνουμε ένας ανοιχτός χώρος για τους πολίτες. Όταν κάποιος θέλει να διαφύγει από τη χώρα του και ζητεί άσυλο, για οποιονδήποτε λόγο και αν οθείται στην πράξη του αυτή και μπαίνει σε ένα καριδότσουφλο, θα χρειάζεται και τη βοήθειά μας. Χρειάζονται λοιπόν διαδικασίες ασύλου, λογικές, ορθολογικές και θα πρέπει και τα κράτη στα οποία φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί στην Νότια Ευρώπη να μην τα αφήσουμε αβοήθητα, όπως είπε και ο Σέρφος νωρίτερα. Θα πρέπει και αυτά τα κράτη λοιπόν να στηρίξουμε. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι οι δημογραφικές εξελίξεις μας υποχρεώνουν να δεχθούμε νέους ανθρώπους, ανθρώπους που έρχονται στον στο άσυλο και που θα θελήσουν να μείνουν στις χώρες μας και όχι να κλείνουμε τις πόρτες. Αυτό το δημογραφικό πρόβλημα μας υποχρεώνει να δεχθούμε και άλλους ανθρώπους ε, από εδώ και μπρος λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Μέλτσερ. Ευχαριστώ πρόεδρο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας ε, λέει με την αποφασή σου ότι είναι απάνθρωπο το σύστημα του ασύλου στην, Ευρω... στην Ελλάδα διότι μπορεί να, διαδικα... να κρατήσουν διαδικασίες ακόμη και πέντε χρόνια. Αλλά δεν να είναι διαδικασίες και στην Ευρώπη ολόκληρη. Χάνονται έγγραφα, ε, χάνονται αιτήσει, ε, κοροϊδεύουν τον υποψήφιο για χορήγηση ασύλου και ακόμα και αν ύστερα από χρόνια παραμονή σε μια χώρα ζητεί για ανθρωπιστικούς λόγους το δικαίωμα της παραμονής. Η Ευρώπη βεβαίω δεν μπορεί να υποδεχθεί στου κόλπους τη όλου του οικονομικού πρόσφυγες. Οι δημοκρατικές εξελίξει λοιπόν και η αναπτυξιακή βοήθεια προς τα κράτη προέλευση αυτών των προσφύγων θα πρέπει να είναι το κύριο μας μέλημα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε ταυτόχρονα και τον ε, ετούντα το άσυλο έτσι ώστε να στηριχθεί σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μέλτσερ, ο κύριος Γιακολίνο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι μεταναστευτικές ροές είναι πολλαπλές. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε ε, μία λύση σε επίπεδο Συμβουλίου. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να διευθετηθεί ένα πολύπλοκο ζήτημα, γιατί η απόφαση σημαίνει ότι δεν θα γίνονται ανούσιες μεταφορές σαν αυτές που ζήσαμε πρόσφατα. Βεβαίως θα πρέπει να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως προϋποτίθεται. Αυτό όμως που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό είναι να μην υπάρχει μία διαφανής ρύθμιση. Και ελπίζω, κυρία Επίτροπε, ότι με ταχύς ρυθμούς θα προωθηθεί σε επίπεδο Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Γιακολίνο. Το λόγο έχει ο κύριος Μέσνερ. Α, με συγχωρείτε, ο κύριος Γκρίσμπεκ. Η κυρία Γκρίσπεκ, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομη θα είναι η ερώτησή μου, διότι η συζήτηση ήταν πολύ ζωηρή και νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επίτροπο πώς θα δεχτεί την εικονοκλαστική ιδέα της ανέγερσης τείχους μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Παρόλο που γνωρίζουμε τις πιέσεις που γνωρίζει αυτή η χώρα και επίσης γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση όταν βρίσκονται σε κέντρα συγκέντρωσης, αλλά η ανέγερση ενός τείχους δεν είναι μια ρεαλιστική λύση, ούτε και σκόπιμη, γιατί γνωρίζουμε ότι συγκυριακά μπορούν να συμβούν πολλά, όπως τώρα βλέπουμε στη Λαμπεντούζα. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε, να αντιμετωπίσουμε συνολικά τις χώρες του Νότου. Θα πρέπει κατεπηγόντως να ξαναδούμε τον κανονισμό του Δουβλίνου για να υπάρχει ανθρώπινη προσέγγιση αυτού του ε, δυσχερού ζητήματο και να δημιουργήσουμε ένα αυθεντικό ε, άσυλο για τους ετούντες στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, ο κύριος Σιλβέστρης έχει το λόγο. Mm, Οι ευρωπαϊκές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπορούν να τεθούν εν αμφιβόλο. Η απόφαση του ΕΔΑΔ μιλά για, μία, για έναν κατεπήγοντα τρόπο σκέψης ως προς αυτά τα ζητήματα. Θα πρέπει λοιπόν να καταρτήσουμε μία ενωτική στρατηγική και οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τάχιστα. Όμως, οι όμορες χώρες είναι χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλο φόρτο και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μία κοινή προσέγγιση. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τις όμορες χώρες να αναλαμβάνουν και το κόστος και το φόρτο. Χρειάζεται επιμερισμός υποχρεώσεων. Και αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει σωστά χωρίς να αμφισβητούμε την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων. Το λόγο έχει η Επίτροπος, η κυρία Μάλστρομ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση. Αυτή η απόφαση είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν υποσκάπτει το σύστημα του Δουβλίνου. Το σύστημα αυτό αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως τονίζει ορισμένα επιμέρους ζητήματα και γι' αυτό θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το σύμφωνο του Δουβλίνου και τον κανονισμό του. Χαίρομαι λοιπόν που προτάθηκε κάτι τέτοιο και χαίρομαι που βλέπετε και την ανάγκη ύπαρξης ενός μηχανισμού κατεπίγουσας ανάγκης. Επίσης, θα πρέπει να ορίσουμε ένα κοινό σύστημα, σύστημα χορήγησης ασύλου. Χαίρομαι για την εργασία μας και θα ήθελα σύντομα με βάση μια έκθεση να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Έχουμε κοινέ αξίες, τηρούμε διεθνείς συμβάσεις και γι' αυτό δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή μεταχείριση των ανθρώπων, θα πρέπει να υπάρχουν αποδοτικά συστήματα έτσι ώστε να μην κρατούνται οι ετούντες για μήνες ή και γιατί αυτό είναι ιδιαίτερα επώδυνο αλλά και δαπανηρό. Για άλλη μια φορά σας ενθαρρύνω μαζί με το Συμβούλιο να συνεχίσετε να εργαζόσαστε. Ως προς την Ελλάδα, η Επιτροπή καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ε, για να βοηθήσει την Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται επί ενός προγράμματος ε, δράσης, όμως υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα, υφέρποντα προβλήματα και ελπίζουμε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και μέσα στα πλαίσια του Frontex, μέσα στα πλαίσια πραγματογνωμοσύνης, διερμηνέων και ούτω καθεξής, να καταδείξουμε αυτή την αλληλεγγύη. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα υφίσταται υπερβολικές πιέσεις αυτή τη στιγμή. Όμως η Ελλάδα φέρει την ε, βασική ευθύνη δεν νομίζω ότι η ανέγερση ενός τείχους επιλύει το πρόβλημα. Υπάρχουν άλλες μεταρρυθμίσεις που είναι πολύ πιο σημαντικές και γι' αυτό ε, εργαζόμαστε με την ΕΑΣ στην Λαβαλέτα για να ενισχύσουμε αυτό το πλαίσιο. Η Τουρκία πρόσφατα δείχνει επικοδομητική στάση μέσα στα πλαίσια επανεισδοχής μετά από 8 χρόνια και ελπίζω στο επόμενο Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα να γίνει αποδεκτό αυτό το πλαίσιο. Ως προς τα αριθμητικά στοιχεία που ζήτησε η κυρία Βίκστρομ για το 9 και το 10 είχαμε 16.000 περίπου αιτήσει προς την Ελλάδα και 12.000 έγιναν αποδεκτές. Όμως τα κράτη-μέλη εκτέλεσαν μόνο 2.251 εκτίσεις, ε, αιτήσεις. Με συγχωρείτε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω άλλη μία φορά για την υποστήριξη της εργασίας μας. Πρόκειται για νομοθετικές ε, πράξεις που βρίσκονται επιτάπητος. Ας εργαστούμε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να καταδείξουμε ότι μπορούμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κοινό σύστημα χορήγησης ασύλου. Ευχαριστούμε την Επίτροπο. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης. Τα άμεσα μέτρα της Ένωσης για την στήριξη της Ιταλίας και των άλλων κρατών μελών που επηρεάζονται από έκτακτη συρροή μεταναστών. Δίνω το λόγο στην Επίτροπο, την κυρία Μάλστρον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ, σα ευχαριστώ για αυτή την εξαιρετικά επίκαιρη συζήτηση. Οφείλουμε ε, να εξετάσουμε την τωρινή κατάσταση.